Καλημέρα σας. Ε, όμως ακόμα οι συνάδελφοι αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόλαβαν να έρθουν γιατί φαίνεται ότι δεν τα πάνε και τόσο καλά όσο θα έπρεπε τα τράμικη γιουνί στο Στασβούργο. Όμως θα αρχίσουμε με την ερώτηση της κυρίας Αντρικένα. Ναι κύριε φίλε. Θα απαντήσετε την υπαριθμόν 20 ερώτηση κυρία Αντρικένε. Μόλις μπορείτε, μόλις είστε έτοιμος, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Όχι, όχι. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που ε, κάναμε αυτή την εσωτερική αλλαγή. Σας ευχαριστούμε για την ευελιξία σας. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ε, τόσο σημαντική και επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Λάιμα Λουσία Αντρικένε, έχουμε να σας πούμε ότι έχουμε υπόψη μας αυτές τις παραβιάσεις των δημοκρατικών διαδικασιών που έχουν καταγγελθεί από μία σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων που έγιναν στις ε, εκλογές τοπικής αυτοδίκης στη Λευκορωσία. Όλα αυτά έχουν αναφερθεί οι λαθροχειρίες, οι απόπειρες νοθείας κλπ. Ή στην καταμέτρηση των ψήφων μας, τα έχει πει η αντιπροσωπεία μας. Έχουν καταγγελθεί όλα αυτά από τις 3 Ιουνίου του 2010 από το Ελληνική Υπηρεσία του ΩΣΑ και θεωρήθηκε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για αποκατάσταση της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση επιδέχεται βελτίωση. Απέχει πολύ από το να θεωρείται επομένως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε και μια αποστολή τον ε, Ιούλιο και θα ευχηθεί προς τις αρχές ότι θα πρέπει να επιφέρουν κάποιες μεταβολές σε πάρα πολλούς τομείς που είναι κλειδιά για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Η Άννη Λευκορωσία ε, έχει σοβαρές προθέσεις προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκλογική νομοθεσία είναι ε, ένας τομέας που θα πρέπει να προσεχθεί. Οπότε, το Μίνσκ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται να συνεργάζεται ούτως ώστε να έχουμε κατά τις επόμενες ε, προεδρικές εκλογές ε, κάποια κατάσταση αποδεκτή. Επίσης θα πρέπει να προσεχθούν και άλλες εκφάνσεις της δημοκρατίας όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε γιατί και εκεί δεν έχουν σημειωθεί βήματα πρόοδου. Κυρία Αντρικένε, λέει ο Πρόεδρος, μήπως έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Αντρικένε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Έχω πρόσθετη ερώτηση. Βλέπουμε ποιε είναι αντιδράσει από παντού σε σχέση με αυτά που είδε στην Λευκορωσία οι Αμερικανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κυρώσεις εις βάρος του, του Μίνσκ. Νομίζω ότι πρόκειται για αντίδραση προς τα όσα έγιναν κατά τις δημοτικές αρχές. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω είναι να μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει όσον αφορά αυτές τις παραβιάσεις της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά όσο γίνονται εκεί. Ο Επίτροπος. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε στο παρελθόν ε, και την πολιτική της συνεργασίας, δοκίμασαμε την πολιτική της απομόνωσης και ειλικρινά καμία από τις δύο αυτές πολιτικές δεν απέδωσε τα όσα εμείς θέλαμε να επιτύχουμε στις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία. Τώρα τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να θέσουμε τα θεμέλια για αυτό που θα ονόμαζα μία συμμετοχή κριτική όμως. Δηλαδή, έχουμε σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα τα περιέγραφα ως ένα πλαίσιο ε, παντός καιρού. Τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας και για τις καλές μέρες και για τις κακές. Ε, έχουμε ένα πλαίσιο λοιπόν ε, που προβλέπει και τον εκδημοκρατισμό και τη σταδιακή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωση στη συνεργασία. Θα προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκεί και βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στη διαδικασία και νομίζω ότι είναι η πιο σωστή απάντηση σε κάτι το οποίο συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι αυτά ε, παρατηρούμε στη Λευκορωσία. Thank you. Mr. Zemker wants to... Ευχαριστώ. Κύριε Ζέμκερ θέλει να κάνει συμπληρωματική ερώτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντηση που μας έδωσε. Αλλά ε, εδώ έχουμε τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, καταλαβαίνω και γνωρίζω ότι ε, σύντομα θα μεταβείτε στη Λευκορωσία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Για τις εθνικές μειονότητες, γιατί, και το λέει και η ερώτηση στο δεύτερο σκέλος, υπάρχουν πολίτες Λευκορώσοι που είναι άλλων εθνοτικών ομάδων, μειονότητες στη χώρα τους. Τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, είναι πολωνικής καταγωγής, αλλά έχουν ε, την ιδιότητα του λευκορώσου πολίτη. Τι γίνεται με αυτούς. Ας, με τις υποτροφίες, ας πούμε. Υποτροφίες για νέους λευκορώσους. Ε, χορηγούνται τέτοιες. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much for this uh, uh, Ευχαριστώ για τη συμπροματική ερώτηση. Υπάρχει ένα τμήμα του προγράμματος που πραγματικά στρέφει την προσοχή του στις ε, διαπροσωπικές επαφές. Ε, να ε, έχουμε ας πούμε, δυνατότητα πρόσβασης από φοιτητέ. Κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα το έχω υπόψη μου στις επαφές που θα έχω εκεί και στις συνομιλίες στο Μίνσκ είναι Ακριβώς όχι τα γενικά ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων, αλλά και τα συγκεκριμένα, τα ειδικά που αφορούν ε, συγκεκριμένες μειονότητε. Και δίδω ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Είχα δε και μία συνάντηση με την κυρία Αντζέλικα Μπόις και άλλους εκπροσώπους της ε, αντιπολίτευσης της χώρας για να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και όχι μόνο την κατάσταση της πολωνικής μειονότητας στη Λευκορωσία, αλλά και με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τη βοηθήσει. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα απομονωμένο, ξεχωριστό ή εκλογικό ή είναι σοβαρό ε, το ζήτημα αυτό, οι σχέσεις ε, του κράτους με τις μειονότητες και θα το θέσω υπόψη του στο Μίνσκ. Ευχαριστώ. Περνούμε στην ερώτηση 18 ε, για τον κύριο Ρέν, 19 για την κυρία Ρέντινγκ και 21 για τον κύριο Ποτότσνικ. Ο κύριος Ποτότσνικ και ο κύριος Μπαρνιέ είναι στο ίδιο τραμ και δεν έχουν φτάσει ακόμα. Α, έφτασαν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρνιέ είναι στο τραμ τότε, καθοδόν. Ε, η ερώτηση παριθμών 18 απευθύνεται στον κύριο Ρεν, όποτε είστε έτοιμος κύριε Επίτροπε. Κράτσα. Είναι της κυρίας Κράτσα η ερώτηση. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα για μια πολύ ουσιαστική σειρά ερωτήσεων γιατί το θέμα της αξιοπιστίας του ευρώ είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους εμάς τους Ευρωπαίους σε αυτή την ε, κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία. Και βεβαίως διότι το ευρώ δεν είναι μόνο μια νομισματική διευθέτηση αλλά και διότι είναι το ένα, το σημαντικότερο αν θέλετε, πολιτικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου η μοίρα του, η αξιοπιστία του, τα όρια του, αυτό έχει επιπτώσει σε, σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να σας πω ότι έχω συντάξει πολύ προσεκτικά μία απάντηση τεσσάρων σελίδων. Ε, ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να συντάξουν την απάντηση αυτή, αλλά αυτό θα σήμαινε, αν τη διάβαζα, 12 ολόκληρα λεπτά. Μπορώ, αν θέλετε, να σας τη δώσω και μπορώ να βάλω και την απάντηση αυτή στην ιστοσελίδα μου, για να μην σπαταλάμε χρόνο. Πράγματι, πρέπει να ληφθούν μέτρα αλλά όσο σημαντικά και είναι αυτά και οι εκστρατείε και οτιδήποτε, το θέμα είναι συγκεκριμένες ενέργειες για να προστατευθεί το ευρώ από τις ε, συστημικές επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε πρόσφατα. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι έχουμε και διεξάγουμε τακτικές ε, έρευνες το Ευρωβαρόμετρο, παραδείγματο χάρη, που ε, γίνεται η έρευνα αυτή σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Στις μελέτες λοιπόν που γίνονται χρησιμοποιούνται όλες οι ευκαιρίες ε, που προσφέρονται για να ε, μεταφερθούν προς τα έξω τα μέτρα για το ευρώ, για την ε, Ευρωπαϊκή, για την Νομισματική Ένωση. Το κοινό λοιπόν, η κοινή γνώμη μπορεί να καταφύγει σε ιστοσελίδες, σε δημοσιεύσεις, σε ενημερωτικά δελτία και σε πολλά άλλα δίκτυα σε φορείς χάραξη πολιτικής, στα συνδικάτα, στις ενώσεις εργοδοτών. Όλα αυτά λοιπόν αν θέλετε για μας είναι μέτρα και ε, πράξεις συνεργασίας με τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουμε την αγωνία μας για το ευρώ. Όσον αφορά τώρα στις πολιτικές οι οποίες βεβαίως βρίσκονται στην ουσία του θέματος αναφέρομαι στο δεύτερο σκέλος ε, της ερώτησης της κυρίας Κράτσα, δηλαδή ποια συγκεκριμένα μέτρα προβλέπετε για την βελτίωση της αξιοπιστίας ε, του ευρώ. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τρία πράγματα. Πρώτον, αποφασίσαμε να συστήσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης τάξη της τάξης των 500 δις ευρώ. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το πακέτο προς την Ελλάδα. Αυτό το μέτρο βοήθησε στο να αναχαιτιστεί η θάμνο πυρκαγιά πριν μετατραπεί σε δάσο πυρκαγιά και κάψει ολόκληρη την Ευρώπη. Εργαστήκαμε λοιπόν πολύ σκληρά για την ε, σταθερότητα του ευρώ. Δεύτερον, τα κρατη έχουν αναλάβει πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Μάλιστα, ε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή λαμβάνονται διάφορα μέτρα εξυγίανσης έτσι ώστε να επανέλθει η αξιοπιστία του ευρώ και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλα αυτά βέβαια ε, τα πράττουμε πολύ προσεκτικά, συνετά και επίσης ε, και με ένα συντονισμένο και διαφοροποιημένο τρόπο έτσι ώστε οι χώρες που έχουν ελάχιστα περιθώρια να επιταχύνουν τη δημοσιονομική τους εξυγίανση, παραδείγματος χάρη Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και πολλές άλλες χώρες και άλλες χώρες οι χώρες εκείνες που έχουν κάποιο περιθώριο στα δημοσιονομικά τους από του χρόνου μπορούν να ξεκινήσουν με την εξυγίανση για να μην καταπνίξουμε την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη που έχει δρομολογηθεί. Έχουμε 15 διαδικασίες ε, αντιμετώπισης του ελλείμματος. Οι στρατηγικές των κρατών μελών ε, για την εξυγένση των δημοσιονομικών τους βρίσκονται σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των ελλημάτων. Και όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι η οικονομική διακυβέρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του ευρώ και εδώ θέλω να πω ότι προσβλέπω στην υποστήριξή σας όταν θα ψηφίσετε για την Ευρώπη του 2020 και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης που είναι απαραίτητη για να πείσουμε το Συμβούλιο και τα κρατημέλη για να παραμείνουμε με τον ίδιο ρυθμό έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, αυστηρά συστήματα ε, εποπτείας ε, και συντονισμό προγράμματα που θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις αρχές του επόμενου έτους. Η κυρία Κράτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και την ευκαιρία που δώσατε να θυμηθούμε όλη την πολιτική για την στήριξη του ενιαίου νομίσματος και την ε, επιβίωση της Ευρωζώνης το πνεύμα της ερώτησής μου ήταν περισσότερο στην επικοινωνία που πρέπει να κάνουμε διότι αυτά τα τεχνικά θέματα και τα πρωτόγνωρα στην ε, οικονομική ζωή της Ευρώπης οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν και δεν τα συμμερίζονται και υπάρχει κίνδυνος να αισθάνονται ότι η στήριξη του ευρώ έχει ένα κόστος και όχι σίγουρο μέλλον. Σε αυτό δεν συμβάλλουν και τα σενάρια και οι απειλές για έξοδο από το ενιαίο νόμισμα κάποιων χωρών. πιστεύω είναι μια συνυπευθυνότητα των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων να στηρίξουν αυτό το επίτευγμα που είναι το ευρώ αλλά η κοινή γνώμη έχει ανάγκη κάποιων υποστηρικτικών μέτρων που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δημοσιονομική προσαρμογή των χωρών τους. σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την επιχειρηματολογία σας και όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ευρώ να θεωρηθεί ως ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο άσκησης πολιτικής για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτήν την βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε για την Ευρώπη και ταυτόχρονα όμως από την άλλη μεριά να το θεωρήσουμε και ένα σύμβολο, ένα, ένα μέσον για να έρθουν πιο κοντά οι Ευρωπαίοι στον άλλο για να μπορέσουμε να χτίσουμε όλοι μαζί τον ευρωπαϊκό οίκο, όπως το θέλουμε. Και με αυτά σχετίζονται και ανακοινώσει μα σε σχέση με τα όσα θέλουμε να κάνουμε, με τα όσα έχουμε προγραμματίσει για τον πρώτο ήμιση του ενεστώτα έτου. Έχουμε και αυτή την ε, ενημερωτική εκστρατεία όσον αφορά ποια είναι τα πλεονεκτήματα ε, στις 10 αυτές χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, Αυστρία, η Φιλανδία, η Μάλτα, Βέλγιο και έχουμε επίσης ε, οργανώσει το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελών, έγινε πριν από δύο εβδομάδες και είχε ως κεντρικό θέμα ε, τα χρηματοοικονομικά ζητήματα της εποχής μας και είχαμε πάνω από χίλιους οι οποίοι ε, Επίση, φυσικά και ήταν ευρύτατη η δημοσιότητα που του προσέδωσαν αυτού του φόρουμ τα μη μη έψιλον. Ε. Και έτσι ελπίζουμε ότι τους διαμορφωτές της γνώμη τους αγγίξαμε και θέλουν απολυστικό αποτέλεσμα μέσω των δημοσιευμάτων του για το φόρουμ. Θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμίσω τις δραστηριότητες μας σχετικά αλλά νομίζω ότι θα αποκομίσουν τα καλύτερα τα αποτελέσματα αν μπορούμε να έχουμε τις ορθές, δόκιμες πολιτικές και να έχουμε τις επίσης πιο σωστές συνοριτικές εκστρατείες ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ο κόσμος είναι καλά ενημερωμένος. Από τα 12 να δουλεύω, πουλάγα ανταλλακτικά. Και ανέκαθεν είχα ξεκάθαρη αντίληψη και φιλοσοφία ότι θα πρέπει να θέτει σε εμπορία το σωστό προϊόν για να πετύχει. Άρα χρειαζόμαστε και εμείς στερε σωστέ πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μια εκστρατεία για να τι προωθούμε ε, σωστή και έτσι να κρατήσουμε το, το μυαλό και την καρδιά του κόσμου. Uh, Υπάρχουν δύο πρόσθετε ερωτήσει, αλλά επιτρέψτε να πω, κύριε Επίτροπε, λέει ο ότι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο παρατηρήσατε, ότι οι συνεργάτε σα σα δώσανε μια επεξήγηση 12 σελίδων και το ανεβάσετε στο website. Ίσως επ' αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε. Πρόκειται για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι ένα τέτοιο σημαντικό θέμα και ερώτημα αξίζει να έχει πλήρη, εκτεταμένη απάντηση και κάλυψη. Αλλά όμω την ώρα των ερωτήσεων δεν έχουμε χρόνο για το τόσο, τόσο πλήρη απαντήσει και πλήρη κάλυψη. ίσω επομένω θα πρέπει η εγγράφο να υποβάλλετε την απάντησή σα για να συμπληρώσετε τόσο θέλετε να πείτε. Να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε. Ο κύριο Κοντή τώρα έχει το λόγο για συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, άκουσα με πολύ προσοχή την απάντησή σας πιστεύω δεν γνωρίζω αν το υπόμνημα που αναφέρατε των δώδεκα σελίδων περιλαμβάνει απάντηση και σε ένα σκέλος που αναφέρεται η ερώτηση της συναδέλφου σχετικά με την ένταξη νέων χωρών στην ευρωζώνη ποια είναι η προοπτική. αφού σας πω ότι γνωρίζω, γνωρίζετε ότι το νέο μέλος είναι η εσθονία αυτό που παρατηρούμε είναι προκειμένου αυτές οι χώρες να μπουν στη ζώνη του ευρώ εφαρμόζουν σκληρά προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης με συνέπεια σήμερα η εσθονία να έχει δραστικές περικοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων η ανεργία να έχει φτάσει στο 20%, η ανεργία των νέων πολλαπλάσια. και το ερώτημά μου είναι αυτή η εικόνα ενός προθαλάμου για, ε, για την ευρωζώνη για το ευρώ είναι ελκυστική είναι αξιόπιστη δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω βιωσιμότητας. ευχαριστώ πολύ. Commissioner. Thank you, Σας ευχαριστώ, αξιότιμη κύριε Βουλευτά, για την ερώτηση αυτή. Ο λόγος για τον οποίο η Εσθονία αναγκάστηκε να επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι κατά κύριο λόγο το ευρώ, αλλά το γεγονός ότι η οικονομία της αντιμετώπισε πάρα πολύ σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, όπως όλοι μας άλλωστε. Και αποτελματώθηκε η μεγέθυνση της οικονομίας και μάλιστα ήταν σε ύφαση. Και τα δημόσια οικονομικά της δεν ήταν πλέον βιώσιμα. 7,2% 75 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με οικονομικούς και μόνο όρους ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει αυτή την ατραπό για να ε, προχωρήσει προς τη σταθεροποίηση των πολιτικών της για να είναι βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Η απόφαση ελήφθη δημοκρατικά ε, στη Βουλή της Εστονίας και ε, είναι η πολιτική που ακολουθεί η χώρα με επιτυχία θα έλεγα. Ο κύριος Παλέτσκης, παρακαλώ για τις ε, συμπροματικές ερωτήσεις. Όχι πάνω από 30 δεύτερα. Είτε είστε συντάκτης ερώτησης, είτε όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο αδύναμος κρίκος στην Ευρωζώνη είναι η Ελλάδα. Δύο μήνες χρειαστήκαμε για να βρούμε ένα μηχανισμό πακέτο στήριξης για την Ελλάδα. Η καθυστέρηση ε, είναι κατά κύριο λόγο κάτι το οποίο οφείλεται στη Γερμανία και μας κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αφήστε δε που υπονόμευσε και το ευρώ ως νόμισμα αυτό καθ' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι βήματα θα πάρει στο μέλλον για να μην έχουμε τέτοιου είδους καθυστερήσεις. I do Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το παιχνίδι απόδοσης ευθυνών. Η δική μου άποψη είναι ότι η πολιτική και κυρίως η οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα πολιτικής βούλησης, όχι όμως μόνο αυτό, είναι και η τέχνη του εφικτού. Αυτή λοιπόν την ε, φορά κάποια στιγμή κατέστη δυνατό εφικτό να ε, προσφερθεί συντονισμένη οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα και αργότερα κατέστη δυνατό να συσταθεί ο μηχανισμός ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Τώρα λοιπόν το σύστημα λειτουργεί σε σχέση με την Ελλάδα. Δόθηκε η πρώτη δόση, 20 δις ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εστάλησαν μέσα Μαΐου. Η Ελλάδα εφαρμόζει ένα κοινό πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τηρεί το ε, μνημόνιο συνεννόησης. Εξάλλου, αποφασίστηκε να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός οικονομικής σταθερότητας ο οποίος θα είναι το κοινοτικό εκείνο όργανο που θα ανέρχεται σε 60 δις ευρώ, ένα εργαλείο 60 δις ευρώ. Αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως εγγύηση πιστώσεων και αυτά τα χρήματα, αυτό το ποσό ε, μπορεί να εκταμιευθεί εφόσον πραγματικά είναι απαραίτητο. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια ειδική ρύθμιση, η διακυβερνητική που και αυτή αποκαλείται ε, οικονομική σταθερότητα. θα ανέρχεται σε 400 δις ευρώ, κατά 90% θα ε, χρηματοδοτείται με βάση τα δικά μας κριτήρια μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και μετά θα μπορεί να ε, θα καταστεί δυνατόν να εκταμιεύονται κονδύλια. Εάν λοιπόν οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα πιεστικές, έχουμε αυτούς τους δύο μηχανισμούς που θα μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι εξή. Βεβαίω με τον τρόπο αυτό μόνο κερδίζουμε χρόνο. Το θέμα είναι η ουσία ότι πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει μια ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση στην Ευρώπη, ε, κάτι το οποίο δεν έγινε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πάμε τώρα στην ερώτηση παριθμών 19. Η κυρία Ρέντινγκ ίσως μπορεί να έρθει μπροστά για να απαντήσει. Ερώτηση υπευλήθη από την κυρία Μαγκίνες. Κέλλη, επίσης. Ο κύριος Κέλλη. Αντί για την κυρία Μαγκίνες θα υποβάλει την συμπληρωματική ερώτηση. Και όταν είστε έτοιμοι κυρία έχετε το λόγο. Well, President, um, I would like... Η Επίτροπος. Στην προφορική ερώτηση Μαγκίνες έχω να πω το εξής, Πρόεδρε. Αν και η αρμοδιότητα αυτών των υπηρεσιών είναι εθνική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστω να βοηθήσει προωθώντα το δικαίωμα των ε, αναπήρων να μπορούν να ζήσουν ε, αυτάρκες, ανεξάρτητοι. Και επόμενε έτσι να έχουμε αυτή την ε, εναλλακτική εκτός των οικοτροφίων και άλλων ιδρυμάτων, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να χαράξει μια στρατηγική 2010-2020 και έτσι να υπάρχει με συνέπεια ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική που έχουμε αποφασίσει για να καλύψουμε τους ε, αναπήρους ούτως ώστε να μπορούν να ζήσουν, ξέρετε. Να βγουν από τα οικοτροφία και τα άλλα ιδρύματα και τα σχετικά συστήματα. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μένους πόρους από τα διαστατικά ταμεία. Βεβαίω σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε προτεραιότητα, αλλά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε από αυτού με τα κράτη-μέλη για άριστε πρακτικέ, καθημερινέ γραμμέ, θα δώσουμε για να δούμε πώ θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα, ούτω ώστε να αποκτήσουν τα άτομα αυτονομία και ανεξαρτησία. Επίση θα πρέπει να μνημονεύσουμε εδώ τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, γιατί και έτσι μπορούμε να άρουμε του φραγμού που υπάρχουν όσον αφορά τη, τη, τη συμμετοχή των ε, αναπήρων ε, στην κοινωνία επίσης ώρες. Και το Κοινωνικό επίσης μπορεί να χρηματοδοτήσει συμβουλές, κατάρτιση που να είναι προσαρμοσμένε στι ανάγκε αυτών των ε, ανθρώπων, να παρενταχθούν στην κοινωνία, να μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορου τομεί επαγγελματικού βίου, στην οικονομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, να προωθηθεί για αυτά τα πρόσωπα και επίσης και μια εκστρατεία ενημέρωση συνειδητοποίηση για να μην έχουμε δυσμενεί διακρίσεις βάρος του. Επίσης μπορούμε να οργανώσουμε κατάρτιση, επανακατάρτιση προσωπικού, ούτω ώστε να έχουμε αυτή τη μετάβαση από τα ιδρύματα σε, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης γειτονιά και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επομένω την αντίστοιχη υποδομή για να μπορέσουν αυτέ οι υπηρεσίε να, να παρέχονται. Επίση, για όλα αυτά έχουμε μία δέσμη μέτρων για να αξιοποιηθούν τα διορθωτικά ταμεία και να αρθούν οι δεσμενές διακρίσεις βάρος των αναπήρων. Αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν την διαχείριση των ε, αρμοδίων οργάνων για να υλοποιήσουν αυτή μας την πολιτική, να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της και τα σχετικά προγράμματα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αλλά τώρα ο κύριο Σκελή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και η κυρία Επίτροπε, εκ μέρου τη κυρία Μαγκίνε, υπέβαλε την ερώτηση. Έχω να σα ευχαριστήσω για αυτήν σα την πλήρη άρτια. Απάντηση έχω δύο συμπληρωματικέ σύντομε ερωτήσει. Πρώτα-πρώτα, πρόκειται να κάνετε κάτι όσον αφορά εκείνου που χρησιμοποίησαν κακός. Με τον τρόπο του πόρους από τα ταμεία όσον αφορά κάποιες εγκαταστάσεις που προορίζονται για τους αναπήρους δεύτερον. Πόσο σύντομα μπορούμε να άρουμε τα κακό κείμενα σε σχέση με τους αναπήρους ή στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Όταν υπάρχουν καταχρήσεις των διαρθρωτικών πόρων, γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επεμβαίνει αλλά υπάρχει βεβαίως η πρωτογενής υποχρέωση και ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη σωστή εκτέλεση της εκάστοτε πολιτικής και να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας εκείνων που ε, είναι μακροχρόνια εισαγμένοι σε ιδρύματα. Το θέμα είναι τώρα αν τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να να με διαφορετικό τρόπο. Εμείς ε, πρέπει να έχουμε δικαίωμα κυρία, Γνωρίζετε ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα στα διαρθρωτικά ταμεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Εναπόκειται όμως στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να διαχειρίζονται από εκεί και πέρα τα προγράμματα και να τα εκτελούν και να τα εφαρμόζουν επιλέγοντας έργα και project. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχουμε δικαίωμα βέτο εμείς, συνεργαζόμαστε ήδη με τα κράτη-μέλη για να αλλάξουμε ε, την πολιτική ε, στα κράτη-μέλη. Παράδειγμα, με τη βουλγαρική κυβέρνηση. όπου επί μία διετία συνεργαστήκαμε για να μην χρησιμοποιεί τα κονδύλια ε, το κράτος ε, σε ιδρύματα με τροφίμους, Δηλαδή να μην ε, δημιουργεί νέα ιδρύματα, ε, γιατί ο στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση, η έξοδος των αναπήρων από τα ιδρύματα. Thank you. Um, I've Ευχαριστώ. Δύο συμπληρωματικές. Ο κύριος Κούρσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για να ευχαριστήσω την κυρία Πίτροπο για την απάντησή της ε, και την προσήλωσή της στην υπόθεση των ατόμων με αναπηρία. Έχω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις εγώ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των διευθυντικών ταμείων, είπατε όντως ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη τίθεται. Στο παρελθόν, ε, επί κομμουνιστικών καθεστώτων, ε, το κράτος είχε κατάσχει ε, διάφορα ανάκτορα για να τα κάνει ιδρύματα στα οποία στέγαζε αναπήρους. Και χρησιμοποίησαν τα διαρθρωτικά ταμεία τώρα για να ε, ανακαινήσουν τα ανάκτορα αυτά, έβγαλαν τους τροφίμους από τα ιδρύματα και ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει εκεί. Υπάρχει καμιά ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για ε, αξιοποίηση ε, αυτών σε επίπεδο κτήματα αγοράς, τουρισμού, θέσεων απασχόλησης. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα παλάτια που έχουν ανακαινιστεί. Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά ότι η αλλαγή καθεστώτος ε, σημαίνει και αλλαγή του τρόπου προσέγγισης της ε, πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά το παρελθόν. Βεβαίως, εναπόκειται στις κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για να δουν α, ε, πώς θα αντιμετωπίσουν τους θεσμούς τους κατά πόσον επιθυμούν να ανακαινήσουν ε, την ε, περιουσία τους ή όχι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όσον αφορά την αποϊδρυματοποίηση, το να μπουν ε, οι, τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία και να μην παραμείνουν σε αυτά τα ιδρύματα, εμείς προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε το προσωπικό της Κομισιόν, το οποίο μεριμνά για τις συζητήσεις ε, με τα κράτη-μέλη σχετικά με τα θέματα αυτά. Στις 29 Απριλίου η Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειών ε, διοργάνωσε ένα σεμινάριο με την επικεφαλίδα. Θα το αποκαλούσατε αυτό σπίτι σας. Και εκεί παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές του θέματος. Έτσι λοιπόν οι δικοί μας οι συνεργάτες γνωρίζουν πολύ καλά ποια πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ώστε στην επαφή με τις διοικήσεις των κρατών μελών να καταβληθούν προσπάθειες για να αλλάξει η νοοτροπία. Εξάλλου υπήρξε και πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, η Περιφερειακής Πολιτικής και, και την άλλη, τη Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ε, τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να εξυπηρετήσουν και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την ανακαίνιση των σπιτιών αλλά και για να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας στις εν λόγω περιοχές άλλη συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Χουντή παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας θέσω ένα πολύ επίκαιρο πιστεύω και συγκεκριμένο θέμα. Στη χώρα μου, στην Ελλάδα και ενδεχομένως σε άλλες χώρες, λόγω των προγραμμάτων λιτότητας περικόπτονται κοινωνικές δαπάνες και πολλές φορές σταματάει η χρηματοδότηση κέντρων και ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ανάπηρους. Έχω μπροστά μου ένα τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο, με ένα μοναδικό κέντρο που προσφέρει υπηρεσίε σε άτομα και κυρίω παιδιά που έχουν προβλήματα όραση και άλλη αναπηρία 50 παιδιά αφέθηκαν στην τύχη του λόγω έλλειψη χρημάτων. Σα ερωτώ, αυτά τα 50 παιδιά μπορούν να ελπίζουν ότι αυτό το ίδρυμα θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. It is ε, very είναι σαφέστατο ότι στην κοινωνική πολιτική τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για να διοργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους, το καθένα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και το ποιοτικό έλεγχο σε συστήματα και ιδρύματα που παρέχουν μακροχρόνια φροντίδα και περίθελψη. Εμείς δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε εκεί. Και βεβαίως ε, για να αλλάξει την πολιτική του, της μία κυβέρνηση, ε, εκείνη είναι αρμόδια. Εμείς μόνο γενικά μέτρα μπορούμε να οθήσουμε προς μία κατεύθυνση, μία κυβέρνηση να φροντίζει τον πληθυσμό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μεταξύ άλλων, ε, καταρτίζει προσωπικό και βοηθάει ε, σε καλύτερη περίθαλψη και φροντίδα. Αλλά τις βασικές αποφάσεις αν θα παρέχεται αυτή ε, η ε, ε, υπηρεσία είναι των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και απαντήσατε. Με χαρά βλέπω ότι κατέφθασε και ο κύριος Μπαρνιέ. Επόμενη ερώτηση είναι για τον κύριο Ποτότσνικ. 21 του κυρίου Ντέιβις. Όποτε μπορείτε κύριε Ποτόσνη, καθίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα κύριε Ντέιβις. Η ερώτησή σας θέτει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις. Όντω στην Κοπεχάγη ήταν απογοητευτικέ οι εξελίξει και τα αποτελέσματα για το περιβάλλον και στην ε, Ντόχα για το ε, εμπόδιο, συγγνώμη, το εμπόριο ε, απειλουμένων ειδών. Σάιτες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν ξέρω κατά, για το μέλλον μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Είναι πολλαπλοί οι λόγοι ε, που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις τις διεθνείς ε, διασκέψεις και θα πρέπει ε, να αναλυθούν μία-μία οι καταστάσεις. Ξέρετε, 27 κρατημέλη είναι δύσκολο να βρουν μία θέση. 500 εκατομμύρια πολίτες να έχουν την ίδια θέση σε περίπλοκα θέματα, σε διεθνείς διαπραγματεύσεις με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, και για τα δύο, και για τη κλιματική αλλαγή και για τις σάιτες, καταλήξαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή γραμμή και είχαμε πολλές δραστηριότητες και προς ε, την κατεύθυνση των διεθνών εταίρων. Πάνω από έξι μήνες πριν τη συνεδρίαση είχαμε καταλήξει σε ε, θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη απανταχού της γης ε, προχώρησαν σε προτάσεις για τις καρχαρίες, τις τίγρης και άλλα απειλούμενα είδη. Αναγνωρίζω όμως ότι για τον ερυθρό τόνο δυστυχώς δεν καταφέραμε να έχουμε τέτοια μεγάλη επιτυχία. Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να δρά καλύτερα στο εσωτερικό της ΣΑΙΤΕΣ μόλις ε, γίνει πλήρες μέρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα εντείνει τις προσπάθειές της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσει τρίτες χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμα να ακυρώσουν τη σύμβαση και την αντίστοιχη ε, τροπολογία για να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προσυπογράψει και να γίνει μέρο. Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτίωσε το συντονισμό της διπλωματικής ε, δράσης και των διπλωματικών πηγών της σε όλο τον κόσμο. Πριν την Κοπεχάγη προετοιμάσαμε μια κοινή θέση, την παρουσιάσαμε παντού και καθ' όλη τη διάρκεια της διάσκεψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε ε, διαβήματα τύπου Τρόικα σε 40 χώρες με κοινέ αποστολές ε, και αυτός επίσης και σε πολλές ε, διμερείς και πολυμερείς επαφές. Οι διαπραγματευτικές ομάδες ε, συζήτησαν ε, με επισκέψεις σε τρίτες χώρες αυτά τα θέματα. Τώρα, πέρα από την Κοπεχάγη και την Τόχα, θα πρέπει να πούμε το εξής. Ένα από του βασικούς στόχου της συνδέξη τη είναι να ενισχυθεί η φωνή της Ένωσης στον κόσμο. Η εφαρμογή τώρα λοιπόν τη συνθήκη τη Αβώνα θα ενισχύσει τη διεθνή μα παρουσία και εκπροσώπηση. Υπό την έννοια αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να ε, εκπροσωπεί προ τα έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που θεωρεί σκόπιμο το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμβάσεις, προβλέπει η συνθήκη να δοθεί εντολή στο Συμβούλιο για θέματα που είναι της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Συμβούλιο μπορεί να ε, δώσει και διαπραγματευτική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αμέσω και πλήρω να συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια και όλα τα στάδια τη διαδικασία. Αυτό τον καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητάει με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη την εφαρμογή του πλαισίου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω επαγρυπνεί ε, να ε, έχει αποτελέσματα και σωστά να εφαρμόζεται η συνθήκη της για να έχουμε ενωμένη φωνή προς τα έξω σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της συνθήκης της Αβώνας τελικά θα αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή. Κάτι που σίγουρα δεν ήταν στο πνεύμα της συνθήκης της Αβώνας. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διοργάνωσής της, της δάσης σε παγκόσμιες διαπραγματεύσεις και για το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για το θέμα. Um, Ο Επίτροπος και εγώ συμφωνούμε ως προς τους στόχους και στηρίζω την Επιτροπή στην, μάχη της με το Συμβούλιο. Όμως ε, βλέπουμε ε, τους Ιάπωνες να πηγαίνουν από, τη, από είναι ένα σημείο στο άλλο ε, φέροντας χρυσό. Εσείς λέτε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι διπλωματικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι είδου συναντήσεις θα έχετε με την κυρία Άστον για να συζητήσετε το πώς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μπορεί να υπαχθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των ε, διπλωματικών δυνατοτήτων μας. Κοιτάξτε, Όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση που κάνατε, εγώ ε, δεν έχω συναντηθεί με την κυρία Κάθη Άστον για να συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές. Ε, όσον αφορά τον ε, τόνο, ερυθρό, ε, πιστεύω ότι η άποψη της Επιτροπής δυστυχώς εγκρίθηκε καθυστερημένα. Και δεύτερον πιστεύω ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο ήταν αυτή που έγινε ε, τελευταία σε επίπεδο κορεπέρ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε ένα μάθημα από αυτή την εμπειρία, αλλά πολύ σωστά επισημάνατε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεργαστούμε και όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, κατά το μέγιστο τρόπο την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πολύ ωραία. Πάμε στην ερώτηση υπαριθμών 22 του κυρίου Γιώργινσον και Αποκινούμε την κυρία Χολ. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, η κυρία Χολ και ο κύριος ε, Γιόργενσεν υπέβαλαν αυτήν την ερώτηση. Η Κομισιόν γνωρίζει μια σειρά μελετών που αφορούν ε, στη συνδυασμένη δράση διαφόρων χημικών ουσιών. Κυρίως στο τέλος του 2009 οι αρχές της Δανίας δημοσίευσαν τα αποτελέσματα από μία σειρά μελέτες που εξέτασαν τις ε, σορευτικές, ε, τη σορευτική επίδραση ε, χημικών ουσιών ενδοκρινικής διαταραχής σε νέους άνδρες και γυναίκες. Η ιδανική αυτή μελέτη οδήγησε στο να εγκριθούν τα αποτελέσματα του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο του 2009 και εκεί η Κομισιόν εκλήθη να εξετάσει ακριβώς το θέμα της ενδοκρινικής διαταραχής να αντιμετωπίσει γενικότερα το πρόβλημα πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι σωρευτικές δράσεις των χημικών ουσιών. Ως προς την ουσία αυτών αυτή τη σωρευτική δράση των χημικών ουσιών, η Κομισιόν πρόσφατα μέσω διαδικτύου παρουσίασε μια τελευταία μελέτη ε, όσον αφορά στο μείγμα της τοξικότητας, αποτέλεσμα διετούς μελέτης. Η Κομισιόν τώρα ε, θέλει να διαβουλευθεί με τους άμεσα εμπλεκόμενους και επίσης έχει υποβάλει και ένα επίσημο αίτημα ως προς το μείγμα της ε, τοξικότητας. Αυτό το έχει υποβάλει ε, στην Επιστημονική Επιτροπή που ασχολείται με τον αντιπισμό κινδύνων και με άλλη επιστροπή που ασχολείται με την κατανάλωση. Η Κομισιόν το αργότερο το 2012 με βάση αυτή τη μελέτη και τις διαδικασίες διαβουλεύσεων θα καταλήξει σε μια έκθεση όπου θα αναφέρεται ε, υπάρχουσα νομοθεσία και η ΡΙΤΣ ε, και θα εξετάζει την έκθεση σε διάφορες χημικές ουσίες. Μετά από όλα αυτά θα εξεταστούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, κατευθυντήριες γραμμές και οι μέθοδοι αξιολόγησης. Από τότε λοιπόν που καταρτίστηκε ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1999 για ενδοκρινική διαταραχή, εμείς έχουμε επενδύσει από τον κοινοτικό μας προπολογισμό για να καταλάβουμε καλύτερα τους μηχανισμούς ε, και τις ουσίες που επηρεάζουν τη λειτουργία ε, των ενδοκρινικών συστημάτων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ενδοκρινική διαταραχή στη νομοθεσία που υπάρχει όπως στην οικανισμό REACH παραδείγματο χάρη. Η Κομισιόν εξάλλου έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνείς ε, πρωτοβουλίες δοκιμών που έχουν σχέση με την ενδοκρινική διαταραχή. Και εξάλλου η Κομισιόν παρουσίασε μια μελέτη ε, για τα επιστημονικά απορίσματα ε, να κατατεθούν ε, προτάσεις για τον εντοπισμό ουσιών που έχουν ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες ενδοκρινικής διαταραχής. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί κατά το επόμενο εξάμεινο, του επόμενου έτους. Θα ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα κοινοτική στρατηγική και επίσης ε, θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία τόσο όσον αφορά το ρίτσο όσο και τον ε, σχεδιασμό. Ε, η Κομισιόν λοιπόν βλέπετε ότι γνωρίζει πολύ καλά τη σοβαρότητα των θεμάτων που θίξατε και η Κομισιόν εργάζεται ουσιαστικά για να αντιμετωπίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι εύκολο γιατί μας λείπουν ακόμα πάρα πολλές γνώσεις. Πάντως πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα ε, το οποίο ε, χρήζει της προσοχής μας στο μέλλον. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, η κυρία, ε, ο κύριος Γιώργενσεν θα υποβάλει την ε, πρώτη ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι το 2012 θα καταθέσετε έκθεση για να δείτε κατά πόσον είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Αυτό μπορούμε να το πούμε ήδη τώρα. Όσοι γνωρίζουν τον κανονισμό REACH γνωρίζουν ότι το μείγμα δεν λαμβάνεται υπόψη σε τέτοιου είδους οσίες. Και αυτό είναι σημαντικό. Ιδίως η πρόληψη στις ε, αγορές και σε σχέση με τα παιδιά και τις εγγύους. Μήπως ε, θα πρέπει η Κομισιόν ήδη τώρα ε, να καταθέσει μία αναθεώρηση του ΡΙΤΣ και εκεί ε, να αναφέρεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ε, να λαμβάνεται υπόψη επιπτώσεις από το μείγμα των ε, χημικών ουσιών. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Όπως προείπα, το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν έχουμε τα δεδομένα που χρειάζονται και ακριβώ όπω είπατε, ε, δεσμό από τη συνθήκη ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή τη ε, σόφρονη διαχείριση και τη προφύλαξη. Όμω θα πρέπει να βρούμε τα δεδομένα που υπάρχουν και θα πρέπει όσο γίνεται με επιστημονική τεκμηρίωση να προχωρήσουμε. Επίση, είπαμε ότι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια το 1999 και από τότε έχουμε εκπονήσει 84 μελέτες. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια. Και χθε πάντως μίλησα με τους ε, αρμόδιους συναδέλφους τόσο ώστε να με ενημερώσουν και τελικά αυτό που βγήκε είναι ότι ακόμη δεν έχουμε τη γνώση, την τεκμηρίωση για να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αυτό το μελετούμε και στο μέλλον θα προχωρήσουμε. Κύριε Χόλ, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αλλά ακόμα νιώθω κάποια ματέωση για απογοήτευση, γιατί μίλαμε για 13 χρόνια. 84 μελέτες όλα αυτά τα χρόνια. Τι γίνεται με τα έμβρια ε, που όμως ξέρουμε είναι η πιο ευαίσθητη στόχη αυτών των συνοπιών, αυτών των φαρμάκων ε, έχουν τόσα προβλήματα και είπατε για την αρχή της προφύλαξης αλλά τι σταματά την Επιτροπή από το να κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες όσον αφορά το REACH και να προβεί στις σχετικές απαγορεύσεις Επίτροπος Σας επαναλαμβάνω, αυτό το είπα και προηγουμένως. Όταν μιλούμε για την αρχή της προφύλαξης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς την εφαρμόζουμε σε κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και με αυτή την μελέτη δεν καταφέραμε να έχουμε την σόρευση των γνώσεων που θέλουμε να έχουμε όπως το ίδιο ισχύει για τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Αυτό που θέλω, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Ε, ασχολούμαι προσωπικά ε, έξι μήνες μόνο με αυτό το θέμα και θα θέλω να δω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού των πραγμάτων στο μέλλον. Κύριε Άκη, έχει συμπληρωματική ερώτηση. Εκ. Οι ισχύοντε κανονισμοί επιτρέπουν την φενόλη α και επομένω, ο καταναλωτή καθημερινά εκτίθεται σε αυτή την ουσία που μπαίνει στο σώμα του αυτή ουσία. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα, για τα τρόφιμα για τη φαινόλη α για το ριτς θα ληφθούν αυτά τα οποία αποφασίστηκαν το 2010 για τα μπιμπερό κλπ. Like all the... Ε, ο Επίτροπος ακριβώς όπως ισχύει για κάθε επιστημονική τεκμηρίωση, εάν αυτό που λέτε ισχύει, θα το λάβουμε υπόψη για την εκπόνηση της πολιτικής μας στο μέλλον. Βεβαίως και θα λάβουμε υπόψη και την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, βήμα-βήμα αυξάνουμε την γνώση μας, την ποιότητα των πληροφοριών που έχουμε και σας διαβεβαιώ Μόλις έχουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται, θα ενεργήσουμε. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποτότσνικ. Και περνάμε τώρα στην ερώτηση παρθών 24 του κύριου Σον Κέλλη, ο οποίος αποσιάζει αυτή τη στιγμή, δεν τον βλέπω στο έδρανό του. Αναλαμβάνει κανένα άλλο την ερώτηση αυτή. Ορίστε. Πολύ ωραία. Για την ερώτηση 24 Ποιος θα απαντήσει? Α, ο κύριος Ποτότσνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Οι πλημμύρες Κατέφτασε ο κύριος Κέλλη. Αγαπητέ κύριε Κέλλη, η οδηγία για τις πλημμύρες εγκρίθηκε το 2007 και η διαδικασία μεταφοράς της είναι καθοδόν. Ε, το περασμένο μήνα οι νέες πλημμύρες μας υπενθύμησαν τις σοβαρές συνέπειες των πλημμυρών και τη σημασία ε, της διαχείρισης κινδύνου από πλημμύρες που είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα και η προστασία. Η οδηγία για τις πλημμύρες απαιτεί από όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ε, ε, συνεκτικά και μεγάλα προγράμματα περιορισμού του κινδύνου. Τα κράτη-μέλη και ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση των προγραμμάτων και τα κράτη σε διασυνοριακά προγράμματα διαχείρισης ε, των υδάτων. Οι πρώτες προθεσμίες έχουν ήδη λήξει. Γιατί, πρώτον, η μεταφορά σε εθνικό δίκαιο κανονικά μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί οδηγία. Μέχρι σήμερα 12 κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένες τη Ιρλανδία έχουν ε, σεβαστεί αυτή την προθεσμία. 10 κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα κοινοποιήσει πότε θα μεταφέρουν την οδηγία στην κοινοτική νομοθεσία και 5 κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει μερική μεταφορά της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφύγει επί παραλήψη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση τώρα ε, των κρατών μελών, διοικητικών μέτρων, η προθεσμία έληξε στις 20, μάλλον, 26 ε, Ιουνίου. 23 κράτη-μέλη μεταξύ αυτών και η Ιρλανδία ε, κοινοποίησαν. θα δούμε κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές και η γεωγραφική κάλυψη συνάδει με την οδηγία. Βασικά ορόσημα όμως ε, στην εφαρμογή απέχουν πόρο ακόμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν τα βήματα αυτά που είναι πρώτον. Η διεξαγωγή προληπτικού ο συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου για τις πλημμύρες το 2011 εντοπίζοντας περιοχές που είναι ε, υψηλού κινδύνου για εμφάνιση πλημμυρών. Επίσης να ε, χαρτογραφήσουν τον κίνδυνο των πλημμυρών μέχρι το 2013. Και τρίτον, να προετοιμάσουμε τα πρώτα σχέδια το 2015 για τη διαχείριση των πλημμυρών. Θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην εκπόνηση και να ε, διαβουλεύονται οι χώρες με τους ενδιαφερομένους. Σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία είναι σε καλό δρόμο η εφαρμογή και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι αργεί να εφαρμόσει την οδηγία Ιρλανδία. Η Ιρλανδία κοινοποίησε τη μεταφορά της οδηγίας στην νομοθεσία της και ε, επίσης δήλωσε ότι κάνει τις διοικητικές προσαρμογές. Καλωσορίζουμε επίσης το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας έχει κάνει ήδη ε, πιλωτική και ασκήσεις ετοιμότητας ε, στο Δουβλίνο και ε, στο νότο της χώρας όπου υπάρχει μια μεγάλη λεκάνη ε, απορροής και έχει προετοιμαστεί και ένα σχέδιο και έχει υποβληθεί στη δημόσια συζήτηση. Και η Ελλανδία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθεί πολύτιμη ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ε, για τρόπους ας πούμε αντιμετώπισης ε, ευνηδίων πλημμυρών ε, από ποτάμια, υπερχείληση ποταμών και διάφορα άλλα. Uh, Θα ήθελα, λέει ο Πρόεδρος, ε, να εξετάσουμε από κοινού τις ε, τρεις ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις γιατί θέλω να εξετάσουμε άλλες δύο ερωτήσεις πριν ολοκληρωθεί η ώρα των ερωταπαντήσεων. Κύριε Higgins, θέλετε συμπληρωματική και ο κύριος Χίγκιν. Θα λοιπόν πολύ σύντομο, ε, σεβόμενο του άλλου. Πρώτα απ' όλα, κύριε Επίτροπε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για πολύ λεπτομερή και συνεκτική απάντηση που την εκτιμώ ιδιαίτερα. Και μία μόνο συμπληρωματική. Στην περίπτωση χωρών οι οποίες δεν θα καλύψουν τις ε, προθεσμίες. Η ε, Κομισιόν δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να τους προσφερθεί ε, το Ταμείο Λεγγύης σε περίπτωση πλημμύρας και αυτό αφορά και το παρελθόν και το μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία αίτηση που αφορά το παρελθόν. κύριος Μίτσελ άκουσα αυτά που λέχθησαν σχετικά με την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Εγώ ε, τυχαίνει να ε, ζω κοντά σε μια περιοχή στο Δουβλίνο όπου μικροί ποταμοί μπορούν να προκαλέσουν τεράστια καταστροφή σε πόλεις. Μήπως λοιπόν μπορεί να προετοιμαστεί ένα ενημερωτικό δελτίο όπου θα καθίσταται σαφές να μην μπλοκάρουμε τις, ε, τους δρόμους διέλευσης ε, των μικρών ποταμών αλλά να αφήνονται ελεύθεροι γιατί αυτά είναι πρακτικά μέτρα ε, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Τίκα. Κύριε Πρόεδρε, η πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας σημαίνει μια διοσυνεραιακή λύση των προβλημάτων, των υδρολογική φύση προβλημάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω και επενδύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική για τα εσωτερικά τη ε, ύδατα. Και νομίζω ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση ε, των περιβαλλοντικών θεμάτων και κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Ο κύριος Higgins, ε, γιατί είπαμε τρεις συμπληρωματικές αλλά θα δώσω κατ' εξαίρεση τον ε, λόγο στον κύριο Higgins. Κοιτάξτε, οι Ιρλανδοί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ιρλανδία ήταν ε, η ολιγορία κατά την οικοδόμηση σπιτιών ε, σε περιοχές ε, που πλημμύρισαν και προκλήθηκαν πάρα πολλές ζημιές. Ε, μήπως μπορείτε να είστε σύντομοι γιατί αύριο όπως ξέρετε θα υπάρξει μια συζήτηση για τις πλημμύρες στην Ευρώπη. Θα είμαι λοιπόν σύντομο κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ε, πολλοί από εσά ε, το ανέφεραν αυτό. Υπάρχουν λοιπόν δύο δυνατότητε. Η μία είναι η πρόληψη όταν ε, απευθύνεται κανεί ε, στο Ταμείο Παρέμβαση. Όταν λοιπόν συμβεί μία θεομηνία, υπάρχουν και άλλες δύο δυνατότητες στις οποίες μπορεί κανείς να καταφύγει αναφέρομαι στο Ταμείο Ελληνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βεβαίως ε, διέπεται από σαφείς κανονισμούς, ε, ορίζεται η ζημιά και στην περίπτωση της ε, Ιρλανδίας η ζημιά που προκλήθηκε ήταν κάτω από το κατόφλι, από το όριο. Και η Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει, αξιολογεί αυτήν την αίτηση, γιατί σας είπα ότι είναι κάτω από το ταμείο που προβλέπετε για να ε, ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. Εάν λοιπόν τελικά αναθεωρηθεί η απόφαση, τότε πράγματι ε, θα ε, προσφερθεί η βοήθεια. Δεν πρέπει όμως να μπερδεύουμε τα πράγματα. Το ποιος είναι ο στόχος του ενός και ποιος ο στόχος του άλλου. Επίσης συμφωνώ όσον αφορά αυτό που είπατε για, την, ε, για τις βέλτιστες πρακτικές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προγράμματα διαχείρισης να γίνονται με σωστό τρόπο, να είναι σωστά προετοιμασμένα. Υπάρχει αυτό το διασυνοριακό στοιχείο και εμείς ε, το στηρίζουμε ανεπιφύλακτα ε, σε αυτή την οδηγία υδάτων, στην προσέγγιση τη διασυνοριακή. Να υπάρχει λοιπόν μια ε, διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για να αναζητούν και διασυνοριακές λύσεις. Τέλος, να πω και το εξής. Το 2012 επιθυμούμε να καταθέσουμε ένα σχέδιο σχετικά με τα ύδατα και τη διαχείρισή τους. Και στο σχέδιο αυτό θα υπάρχουν τρία θέματα. Ένα από αυτά, σας το επισημαίνω, είναι η ξηρασία και θέματα που έχουν σχέση με την ξηρασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε όλους και όπως σας είπα αύριο προβλέπεται συζήτηση για τις πλημμύρες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, στην υπαριθμόν 25. Κύριε Ποτότσνικ, έχετε επ' το λόγο. Η ερωτήση σας τη Ρεντβίλη Μουρκουνά. Thank you. Σας ευχαριστώ λέει ο Επίτροπος όντως δυνάμει τη σχετική οδηγία και τη ε, μελέτη αξιολόγηση αντικτύπων, είπαμε ότι οι σχετικέ πληροφορίε θα πρέπει να, να, να, χορηγούνται από τι αρμόδιες αρχέ στον εργολάβο. όμως αυτό δεν έχει οδηγήσει σε μια διαδικασία ε, διαφανή, γιατί υπάρχουν πάρα, πολλά, πάρα πολλέ που τάσει η οδηγία αυτή. Όμως Αυτές οι ρήτρες διασφάλισης υπάρχουν όσον αφορά το, το, το τι ορίζεται ως ελάχιστες πληροφορίες στην ε, περιβαλλοντική εκτίμηση και αυτά τα, τα, τα, τα ορίζει ρητός η ισχύουσα οδηγία, αλλά αυτό ισχύει και όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και με τον κόσμο. Και όλες αυτές οι πληροφορίες από τον εργολάβο θα πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως και επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαβουλεύση και με τον κόσμο. Η ιδέα ακρίβεια των πληροφοριών αυτών είναι δυνατόν να προσληθεί αναπάν σημείο τη διαδρομή διαδικασία των διαπραγματεύσεων πριν ληφθεί η οριστική απόφαση. Τούτο σημαίνει ότι οι αρμόδιε περιβαλλοντικέ ε, αρχέ είναι δυνατόν οι ίδιε με δικά του μέσα να προχωρήσουν ει αξιολόγηση τη ακρίβεια των πληροφοριών ε, σε συνεργασία ή το κάνουν για μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι δυνατόν να υποβάλουν στάσει κατά αυτής της διαδικασίας αν θεωρηθεί ότι οι μελέτες δεν είναι ακριβείς ή ότι δεν είναι δεν συνάδουν αυτές οι αξιολογήσεις με τα όσα επιτάσσει η οδηγία ΕΠΕ και θα πρέπει επομένω να συνεκτιμηθούν αυτές όλες οι πληροφορίες και όλα αυτά είναι προσβάσιμα από τον κόσμο. Όμως πάρα πολύ ευστοχή η ερώτησή σας γιατί με μετά από πάνω, πάνω μία εικοσαετία εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή, βρήκαμε που χρειάζεται να επιφέρουμε κάποιε βελτιώσει. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία ΕΠΕ θα πρέπει να υποστεί αναθεώρηση. Στόχο είναι το να έχουμε ένα νέο κείμενο. Έτσι, να βελτιώσουμε την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την βιοπικιλότητα, την ενεργειακή πολιτική, το περιβάλλον, τις σχετικές ορθωτές προκλήσεις, λάβουμε υπόψη την νομολογία του ΔΕΚ και να προσθέσουμε τις ισχύουσες ε, διαδικασίες στα πλαίσια αυτά. Η ποιότητα των αξιολογήσεων θα, θα είναι στο επίκεντρο ε, του έργου μας, γιατί βεβαίως και επειδή έχει την κατάσταση βελτιώσει, από μια μεριά ο ποιοτικό έλεγχος της ε, ΕΠΕ, των πληροφοριών του εργολάβου και η ίδια αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να περιχαρακωθεί και οι υπηρεσίες μας ήδη άρχισαν να δουλεύουν όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας και περί τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε μια εκτεταμένη διαβούλευση με τον κόσμο, με όλους τους εμπλεκομένους και εσείς επίσης ε, είστε καλοδεχούμενοι να συμμετάσχετε να πείτε τις απόψεις και μόλις έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες τα δεδομένα τότε η Κομισιόν θα δει τι επιλογές υπάρχουν όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας και πώς θα εξασφαλίσουμε το πώς θα είναι αντικειμενικές οι μελέτες αξιολόγησης και κάθε πρόταση θα πρέπει να περάσει από αυτή την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ακόμα δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω πότε θα κατεβάσουμε τις προτάσεις μας, όμως θέλω κατά τη θητεία μου όλα αυτά να τα ξανασυζητήσουμε όσο γίνεται γίνεται αλλά πρώτα πρώτα θα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί για προετοιμασία. Ευχαριστούμε κύριε ο Πρόεδρος. Μας Λένε οι διερμηνείς ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Διαβάζετε γρήγορα. Όμως, έχουμε ακόμα μπροστά μας δουλειά και όλα αυτά που λέτε ε, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα. Τώρα κύριε Μικουλενιάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και για τα κράτη-μέλη αλλά και για άλλους φορείς. Τα έργα υποδομής έχουν σημασία σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε έργα υποδομής ας πούμε για ενεργειακά ε, ζητήματα, αγωγούς, στον αγωγό North Stream, στη Βαλτική θάλασσα. Και είπατε ότι θα πρέπει να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών ε, στη διαδικασία και να λαμβάνονται υπόψη τα μελήματα για ανησυχίες της. Αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν έλαβε υπόψη του τις πληροφορίες που δίνουν ανεξάρτητοι επιστήμονες και μιλούν για τη δυνατότητα και για την ανάγκη να ε, είμαστε ε, ανεξάρτητοι όταν κάνουμε μελέτες ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εσείς τι λέτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετέχει, θα ελέγχει τα κρατημέλη αν κάνουν σωστά τις μελέτες αντικτύπου. Θέλετε να απαντήσετε. Yeah, in essence... Uh, ναι, στην ουσία και πάλι σωστά είναι αυτά που λέτε. Έχετε δίκιο. αν ένα έργο ή μια επένδυση δεν έχει διασυνοριακές επιπτώσεις, είναι σαφής η διαδικασία. Εκεί μπαίνει η επικουρικότητα. Και δεν θα είχα τίποτα άλλο να προσθέσω. Όταν είναι διαφανής η διαδικασία και όλοι έχουν ε, συμμετοχή και άποψη, που κατά τα άλλα ήταν και η πρόθεση της προηγούμενης αναθεώρησης οδηγίας αυτής το 2003, τα πράγματα είναι εντάξει ευθυγραμμίστηκε με τη σύμβαση του Άρχους και βεβαίως η διαδικασία κανονικά θα πρέπει να οδηγεί και να διέπεται από τις αξίες που αναφέρεται. Τα πράγματα περιπλέκονται όντως όταν μιλούμε για διασυνοριακά έργα υποδομής. Αυτό που ζητάει σήμερα η οδηγία στη διασυνοριακή συνεργασία είναι να υπάρχει διαπραγμάτευση ή μάλλον καλύτερα ε, ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης με τους ενδιαφερομένους αυτό πώς γίνεται. Με την ίδια τη σύμβαση ΕΣΠΟ, αλλά μπορούν και τα κράτη-μέλη τα ίδια να συμμετέχουν και εκεί βρίσκει εφαρμογή παρούσα οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειλικρινά, πώς να το πω, έχουμε μάλλον διαδικαστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς να τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες ιδεοδός θα οδηγούσαν σε μια μελέτη αντικτύπου ανεξάρτητη ε, ε, που θα την κάνει πρώτα ο εργολάβος, αν χρειαστεί να την ελέγχει στη συνέχεια ε, το κράτος μέλος και αρμόδιες αρχές κτλ. Αλλά βεβαίως όλα αυτά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Στο πνεύμα της οδηγίας αυτής έχουμε βάλει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι το περιβάλλον λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν γίνεται οποιοδήποτε τέτοιο έργο και οποιαδήποτε επένδυση. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι η δημόσια διαβούλευση γίνεται πάντα με τρόπο διαφανή. Αλλά σωστά τα λέτε κι εσείς ότι μάλλον υπονοείται ότι ε, εκκρεμούν ακόμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση σε ποια κατεύθυνση θα πάει η συζήτηση. Είναι ακόμα ανοιχτή. Τώρα ξεκινάει. Και σίγουρα στο μέλλον θα κοιτάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Thank you. Mr. you asked for... Ευχαριστώ. Κύριε Ζέμκερ, ζήτησε συμπληρωματική ερώτηση, αλλά δοθέντως ότι ήδη ρωτήσατε σήμερα και επειδή έχει προχωρήσει η ώρα δεν θα σας δώσω το λόγο. After the next... Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Και μετά, τέλος, ζητώ συγγνώμη για τους συναδέλφους που ήρθαν για να ακούσουν τι απαντήσει του κυρίου Μπαρνιέ. Θα τι δώσει γραπτό σε όλους σας. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε στις 8.30 για τον απλούστατο λόγο ότι στις 9 ξαναρχίζουν οι διερμηνείς να δουλεύουν και κάποτε πρέπει να φάμε κιόλας. Ε, επόμενη ερώτηση. Okay, fine. I'm used to this. Uh, ναι, ναι, τα ξέρω αυτά, τα έχω συνηθίσει, ωραία. Δεν υπάρχει τρόπος να το αλλάξουμε αυτό. Ε, για λόγους τάξεως, σας παρακαλώ. Πρώτα οι κυρίες. Χάρκιν ε, και μετά η Lady Λάτφορντ. Πρώτα η κυρία Χάρκιν. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη πρόεδρε. Απλώς θέλω να υποβάλω την ερώτηση. γιατί πέντε πήγαν σε έναν επίτροπο και ένα σε άλλον. Μα είναι αυτό θεμητό, είναι δίκαιο. Δεν θα έπρεπε να, καλύτερα να βαλουμε 3 3-3 τρει να, είναι, να είναι πιο ισόρροπη κατανοημένο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποιο είναι ο λόγο που κάνετε αυτή την κατανομή. Ε, όποιο, η προτεραιότητα δόθηκε σε όποιον ε, ρώτησε πρώτο. Ε, Λάτφορτ. Ναι. Και ο άλλος επίτροπος πάει, καμία ερώτηση. And then, and then Ο κύριος Ντάλι τίποτα τον, χάσαμε. Δεν νομίζω ότι έτσι πολύ καλά τα χειριστήκατε και έτσι ε, πάει ο ένας επίτροπος. Δύο, δύο, δύο δεν θα μιλήσουν. Κύριε Χάρμπορ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Παρακαλώ να αναφέρετε εις το Προεδρείο ότι ό,τι ως πρόεδρος εσωτερικής αγοράς δεν μπόρεσα να ακούσω δύο από τους επιτρόπους, τους αρμοδίους για την επιτροπή μου. Γιατί ξέρετε τι ισχύει και εσείς και η γραμματεία όταν άρχισε η συνεδρίασή μας ότι είχαμε συγκεκριμένο περιορισμένο χρόνο στη ε, διάθεσή μας γιατί πρώτα πρώτα μπορούσατε να παρέψετε τι δύο ερωτήσει που συζητήσαμε στην αρχή. Δεν είχαν να κάνουμε κανέναν επιτρόπου του παρόντε, γιατί εδώ πέρα ήρθε κόσμο ακριβώ για αυτού του επιτρόπου. Μπορούσατε εκείνε να τι αφήσετε. Μπα και πρέπει να αλλάξει ο οργανισμό επί του θέματο. Δεύτερον, είναι σαφέ πόσο χρόνο έχουμε. Επομένω, μπορούσατε να μοιράσετε τι ερωτήσει μεταξύ των επιτρόπων που είχαν την καλοσύνη να κάνουν τον κόπο να έρθουν εδώ. Είναι τερατώδες ότι αγνοούμε δύο επιτρόπους που ήρθαν εδώ. Δεν τους δίνουμε καθόλου χρόνο. Εσείς επομένως ως Προεδρεύων, παρακαλώ, εγώ σας το ζητώ ως πρόεδρος της Κοινοβουλικής Επιτροπής να αναφέρετε σχετικό στο Προεδρείο και να πείτε ότι είμαστε έντονα δυσαρεστημένοι διότι ε, η διαδικασία ε, διευθύνεται με τρόπο απαράδεκτο πρόεδρος. Πάντως όλα τα κοινοβούλια δεν προκάνουν όσον αφορά να το ρωτήσουν. Δεν προκάνουν να τελειώσουν. Κύριε Πότστα θα σα δώσω το λόγο. Κύριε Παπαστάμκο, έχετε εσεί το λόγο. Πράζω και εγώ την, ε, την έλλειψη, ε, την ορθολογική έλλειψη κατανομής ε, του χρόνου. Ε, κύριε Πρόεδρε, παράλληλα είχα Επιτροπή Γεωργίας και ψηφοφορίες και άφησα την Επιτροπή και ψηφοφορίες για να είμαι συνεπής την ώρα αυτή του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι προφανές ότι δεν κάνατε σωστή κατανομή του χρόνου μεταξύ των μερών του κοινοβουλευτικού ελέγχου επιτρέπατε συμπληρωματικές ερωτήσεις κατά τρόπο ε, πάρα πολύ ε, ευέλικτο και ε, νομίζω ότι και απέναντι στους επιτρόπους και στον κύριο Μπαρνέ πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Αυτό επιτάσσει η κοινοβουλευτική τάξη και το λέω εσάς κύριε Πρόεδρε που προσωπικά σας εκτιμώ προέρχεστε από τη χώρα όπου καθιδρύθηκε η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία αλλά η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει και τάξεις έχει κανονισμό έχει και αρχές. λυπούμε πάρα πολύ για αυτό που έγινε απόψε. δεν τιμά κανέναν και δεν τιμά το κοινοβούλιο αλλά δεν τιμά και το προεδρείο κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί ήταν απόντες οι επίτροποι μεταξύ άλλων. Ο κύριος ε, Πόσελτ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, από το 1994 συμμετείχα σε όλες τις ώρες των ερωτήσεων. Τέτοιο σκάνδαλο δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι τελείως φυσιολογικό. Όταν μειώνεται ο χρόνος να κόβεται από κάθε επίτροπο κάτι. Την πρώτη ερώτηση του κυρίου Ντάλη έχω εγώ και ήξερα ότι θα έρθει η ερώτησή μου. Τώρα ο κύριος Μπαρόζο είναι στην πολιτική μου ομάδα και εγώ έφυγα πριν από τρία τέταρτα για να έρθω εδώ. Και κάθομαι 45 λεπτά και περιμένω να έρθει η σειρά μου. Θα μπορούσατε να με είχατε ενημερώσει. Πρέπει να πω ότι με αυτή τη διαδικασία δεν συμφωνώ καθόλου. Και παρακαλώ για τον ερωτήσω να μην περικόπτεται. Είναι το σημαντικότερο σαν ένα κοινοβούλιο. Δεν είμαστε μηχανή εδώ για να ψηφίζουμε για το κατεστημένο. Είναι δικαίωμα κάθε μεμονωμένου βουλευτού, στοιχειώδες, από το Βρετανικό κοινοβουλευτισμό τα έχουμε αυτά ε, κληρονομήσει. Όπως σας είπα, τι να κάνουμε σε όλα τα κοινοβούλια ε, όλου του κόσμου οι ρωταπαντήσεις κάπου τελειώνουν και τελειώσανε. Ευχαριστώ. Οι Οδηγίε περί και οικοτόπων και οι δύο δίνουν την απαραίτητη ευελιξία για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συμβατότητα μεταξύ ε, ανάπτυξης της οικονομίας και προστασίας της φύσης. Η νέα νομοθεσία για τη φύση δίνει ένα συνολικό μοντέλο για την προστασία της φύσης ε, επιστημονικό που να εφαρμόζεται ε, με βάση τον νόμο και τα οικοσυστήματα. Το... Και Το δίκτυο Natura είναι από τα σημαντικότερα συστήματα για την προστασία της φύσης και από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιοποικιλότητα είναι βασική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας. Φέτος το Μάρτιο το Συμβούλιο επαναδιατράνωσε ότι αυτά τα προστατευόμενα είδη και βιότοποι είναι εκ των όνων για τη βιοπικιλότητα και θα πρέπει να ε, ολοκληρωθεί το δίκτυο Natura Φύση 2000 το συντομότερο. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση εκτέλεσης και εφαρμογής της νομοθεσίας και η διαδικασία ολοκληρώνεται και στόχος πλέον είναι να βεβαιωθούμε ότι το δίκτυο Φύση 2000 θα τη χάνει καλής διαχείρισης και σωστής χρηματοδότησης για να μπορεί πλήρως να ανταποκρίνεται στους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους είναι ένα μοναδικό εργαλείο. Επιτρέπει την ε, γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλία, τη δασοπονία και δεν καταστρέφει ε, την φυσική μας κληρονομιά. Οι οικότοποι τη Νατούρα ε, δεν είναι χώροι απαγορευμένοι που απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και οικονομική επένδυση είναι ζωντανά τοπία η οικοτοπία αυτή και οι άνθρωποι ε, συμβιούν με τη φύση. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να παγώσουν όλες οι οικονομικές και ανθρώπινες δραστηριότητες εκεί. Το αντίθετο, έχουμε πολλούς ε, οικοτόπους όπως είναι ο Λιμένας της Αμβέρσας που πρόσφατα επισκέφτηκα και έχει σχέση η ερώτησή σας όπου συνεχίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα χέρι με χέρι με την προστασία της φύσης. θα πρέπει από νωρί να συμπεριλαμβάνεται το περιβάλλον στην ανάπτυξη ε, και να τα γνωρίζουν όλοι οι ενδεφερόμενοι για να έχουμε επιτυχή έκβαση όλων των εγχειρημάτων. Ξέρω ότι δεν έχουμε φτάσει στο 2010 στην εκπλήρωση των στόχων μας, θα πρέπει να αξιολογήσουμε για ποιο λόγο δείχθηκαμε στην αποτυχία αυτή, ποιους λόγους και θα πρέπει να δούμε ε, τι πταίει ή τι πταίει και τι βελτιώσεις κανονικά ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται. Η κυρία τα έχετε συμπληρωματική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αυτά ήθελα να ακούσω, γιατί νομίζω ότι όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και όλοι οι οικονομικοί παράγοντες θεωρούν ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτή η οδηγία. Πολύ χαρά που τα άκουσα από εσά και σε ευχαριστώ, Επίτροπε. Πολύ ωραία. Κανοποιημένο, Ναι. Λέει ο Επίτροπος. Άρα όλοι εντάξει. Ευχαριστημένοι. Οπότε διακόπτουμε και τα σε εννέα. Γεια σας.